Therefore we Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε τόσο το καλύτερο. Ε, είμαστε πολύ άσχολοι, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε μέχρι τις 10. Μέχρι τότε, σε μία ώρα δηλαδή, μόλις μία ωρίτσα από τώρα, κάποιοι συνάδελφοι θα βιαστούν να μπουν τα συνηθισμένα, θα κάνουν φασαρία, θα μας ανησυχήσουν και θα μας διώξουν. Θα μας πιέσουν να φύγουμε το πρώτο σημείο της διάταξης. Καταπολέμηση της απάτης είναι το θέμα. Κατά της απάτης που στρέφεται κατά των ε, συμφερόντων των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ποινικού δικαίου. Να υιοθετήσουμε την ημίσια διάταξη να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Και μετά την ευκαιρία θα έχουμε για πρώτη φορά μεικτή συνεδρίαση, κοινή συνεδρίαση. Η Κοντ και η Λίμπε μαζί συνεδριάζουν. Χαιρετίζουμε την παρουσία των μελών της Επιτροπής Κοντ και τον πρόεδρο Τόιντερ, την πρόεδρο Τόιντερ, συμπρόεδρο, τον συμπρόεδρο, για να συζητήσουμε ένα κοινό θέμα. Και συμπεριλαμβάνεται και συνεργασία με την Επιτροπή τη Νομική όσον αφορά κάποια άρθρα του φακέλου την καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω ποινικού δικαίου και ποιος είναι ο νομικός όρος του δημοσίου υπαλλήλου. Να αναφέρω λοιπόν τι διακυβεύεται εδώ και να σας θυμίσω ότι πρέπει να προσέξουμε το χρόνο. Μία ώρα έχουμε. 10 και πρέπει να ψηφίσουμε στις 10, λέει ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας. Τον Ιούλιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για οδηγία. πολέμηση της απάτης μέσω ποινικού δικαίου τίτλους. Ευρωπαϊκός, λοιπόν, Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο εν τη διαμορφώση του. Άθο 325 νομική βάση της συνθήκης. Είναι το άθρο της συνθήκης η νομική βάση εναρμόνιση και ενίσχυση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά τα ποινικά δικήματα που σχετίζονται με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτά τα δικήματα επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συμπεριλαμβάνεται η απάτη, παρεμπόδιση των δημοσίων προμηθειών, διαδικασίες χορηγιών, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματων ε, και ατασταλίες διάφορες και υπεξαιρέσεις. Αποφάσισε έσκυψη των Προέδρων τον Μάιο του 2013 ότι Λίμπε και Κοντ θα εξετάσουν από κοινού το θέμα. Δυνάμει το άρθρο 51 του εσωτερικού κανονισμού. Η νομική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του δημόσιου υπαλλήλου και διατάξει για ενεργητική και παθητική διαφθορά θα εξεταστούν από κοινού με την Κοντ, Γιούρι και Λίμπη βάσει του άρθρου 50. Ξεκινάει η συζήτηση. Η νομική επιτροπή εξέδωσε γνωμοδότηση. Εκεί τίθεται το θέμα κατά πόσο είναι σωστή η νομική βάση του 325 και κατά πόσο θα έπρεπε να είναι το 83, που είναι η νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Καθορίζει τα ποινικά δικήματα και προβλέπει την επιβολή ποινικών κυρώσεων. Ελάχιστε προδιαγραφέ. Έτσι συνοψιστεί η κατάσταση λοιπόν, ως εξή. Αντίθετα με το άρθρο 83, το άρθρο 325 δεν υπόκειται σε κανόνες του, της τροχοπέδης κατεπηγούσης ή emergency break. Αυτό να κάτι επηρεάζει Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η πρόβλεψη. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο πλησιάζει με κοινή προσέγγιση. Περιμένουμε ενημέρωση από το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε την κυρία Λεμπάη που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει απόψεις για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και του συμπρόδρο Μιχαήλ Τόιντερ που είναι παρόν στην αίθουσα κι αυτός. Θα πάρει το λόγο πριν εγώ σαν εισηγητής υπεύθυνος στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών προβώ στα πρώτα σχόλια περί των απόψεων που υπάρχουν για το θέμα που θα ανοίξει το δρόμο ώστε στο προβλέψιμο μέλλον δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία. Κυρία Τόιλερ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ως πρόεδρος της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού επίσης να σας ε, χαιρετήσω θερμά και να σας καλωσορίσω. Βλέπετε εδώ στην αθρώα συμμετοχή ότι το θέμα για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και το συμπεριλάβαμε κατά επανάληψη στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο της δικής μας Επιτροπής αλλά και της Ολομέλειας. Και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως θα θέλαμε να υπάρχει περισσότερη απήχηση στην πολιτική συζήτηση σε σχέση με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τα θέματα που, που ανέφερε ο συνάδελφος Λόπες Αγγιλάρ, δηλαδή η καταπολέμηση της απάτης και η δίωξη ε, ε κατά των περσικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι πολιτικά θέματα μέσα των οποίων μπορεί κανείς να κάνει πηχαίως τίτλους σε εφημερίδες αλλά είναι τομείς ε, και τους οποίους πρέπει να φροντίσουμε εμείς. Ε, και γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν για να κλείξει ένα, καλύψει ένα νομικό κενό. Ε, σε, συνάρτηση με τις διαβουλεύσεις μας, όπου η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να προστατεύσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και καταρχήν ορίζοντάς τα η δική μας εισηγήτρια, Ingeborg Γκρέσλε, κλήθηκε να κάνει μια γνωμοδότηση. Αλλά προηγουμένω θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει. Αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Λόπεθ Αγγιλάρα, αγαπητοί συνάδελφοι των δύο υποτροπών, χθε είχαμε μια εντατική συζήτηση με τον Επίτροπο κύριο Σεμέτα, που κατόπιν δική μου πρωτοβουλία ήρθε σε εμά στην Επιτροπή για να συζητήσουμε και πάλι την ετήσια έκθεση τη Επιτροπή Παρακολούθηση τη Όλαφ. Και στο πλαίσιο αυτό διαπιστώσαμε ότι ε, ε, στο μέχρι τώρα μέχρι προσπάθειες με την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης. Ασφαλώς συμβάλαμε σημαντικά στην ε, καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των άνεμων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διαπιστώσαμε στο πλαίσιο της συζήτησης ότι εδώ προσκρούμε σε κάποια όρια. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο σε δύο τομείς να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Καταρχήν, ε, στο θέμα της ε, εισαγγελία σε, ευρωπαϊκή, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον οικονομικό τομέα και το ζήτημα πώς μπορεί μέσω, κανείς, μέσω του ποινικού δικαίου να βελτιώσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε είναι το θέμα της νομικής βάσης. Και εδώ θα πρέπει εκ των προτέρων να συνεννοηθούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί εδώ στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχαμε μια συζήτηση για τη νομική... υπήρξε μια συζήτηση για τη νομική βάση, αλλά δεν θα ήθελα να προκαταλάβω τα όσα θα πει η συγγήτρια. Χαίρομαι για την κοινή αυτή συνεδρίαση και προτείνω καταρχήν ε, να προωθήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, ούτω ώστε να καταλήξουμε και σε κάποιες ε, αποφάσεις. Από τη δική μας πλευρά, η συνάδελφος κυρία Γκρέσλε ως εισηγήτρια θα πάρει το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω κάποιο σχόλιο να κάνω σαν εισηγητή για την Επιτροπή Ελευθεριών. Uh, να κάνουμε εισαγωγή λοιπόν στο θέμα. Πράγματι, αυτή η εντολή επικεντρώθηκε κατά πολύ στην ανταπόκριση έναντι της οικονομικής και κοινωνικής διαστάσεως της κρίσεως που παραμελήσαμε επί μακρόν. Και ένα από τα σημαντικά βήματα της συνδείξης της Αβώνας ήταν ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά λέγω να θεσπίζει ποινικό δίκαιο. Να γίνει νομοθέτης σε ποινικά θέματα. Νομοθέτης για ποινικά θέματα επαναλαμβάνω. Και ακριβώς είναι από τα μεγαλύτερα βήματα πρόοδου. Αυτό περιλαμβάνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευρύνεται έτσι σημαντικά η εξουσία που έχει το, ο τομέας που έχουμε στον τομέα της ελευθερίας δικαιοσύνης που προβλέπει στη δίκη της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να αποτιμούμε λοιπόν το θέμα και το πόσο σημαντικό είναι ούτε μπορεί να υποτιμάται το μέγεθος της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπολογίζεται ότι βρίσκεται συγκλονιστικά επίπεδα. Δεν θα είμαστε αξιόπιστοι όσον αφορά την καταπολέμηση της οικονομικής και δημοσιονομικής της σηματοστής της κρίσης, εάν δεν είμαστε άντεκτοι στην καταπολέμηση διαφθοράς. Πρέπει να θεσπίσουμε ελάχιστες προδιαγραφές για τις κυρώσεις να καθορίσουμε τα ποινικά δικήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόφλια για τα κράτη-μέλη και κυρώσει είναι από τα σημαντικά θέματα, το ουσιαστικό περιεχόμενο της πρωτοβουλίας. Και είναι γεγονός ότι στο προηγούμενο μέλλον ο... θα πετύχουμε το στόχο όταν θα μπορούμε να έχουμε δικό μας Ευρωπαίους Αγγελέα, όπως το βλέπετε στη συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 86 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σαν πρώτο βήμα όμως αυτή η πρωτοβουλία αρκεί. Διότι καλύπτει τις δυνατότητες θεσπίσεως βασικών προδιαγραφών όσον αφορά τα δικήματα που, και τα εγκλήματα που θα καθοριστούν και κυρώσεις για τα ποινικά δικήματα. Ας συζητήσουμε λοιπόν τους ορισμούς και μετά θα ακούσουμε τον υπεύθυνο εισηγητή της Επιτροπής ΣΚΟΝ, διότι είναι ορμοδιότητά της. Τα οικονομικά συμφέροντα και οι απειλές κατά αυτών και οι βλάβες στις οποίες υπόκειται ο Ευρωπαϊκός Οπολογισμός, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τόνισε ότι σημειώνεται ο ορισμός του άρθρου 2 της προτάσεως διότι αναφέρεται σε εισοδήματα και δαπάνες και έξοδα που καλύπτονται, αποκτώνται ή οφείλονται στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή ή προπολογισμού θεσμικών οργάνων, υπηρεσιών και φορέων. Όμω ο όρο προπολογισμό αμφισβητείται. Συζητείται μεταξύ θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο ορισμό για να αντικατοπτρίζεται το ότι τα οικονομικά συμφέροντα τη Ενώσεω σχετίζονται με όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που διαχειρίζεται η Ένωση ή διαχειρίζεται κάποιο εκ μέρου ενό θεσμικών οργάνων και όλε τι συναλλαγέ, δανεισμό, δανειοληψία, δανειοδοσία. Είναι θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στο φόρο το ΦΠΑ. Φόρο θέμενη αξία. Τόνισε το ελεκτικό συνέδριο ότι φόρο θέμενη αξία και απάτη σε αυτόν το τομέα καλύπτονται από την προτινόμενη οδηγία. Συμφωνεί ότι αυτού του είδους οι απάτες μπορούν να πλήξουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ενώσεως, παρόλο που μεγαλύτερο αντίκτυπο ε, δέχονται τα κράτη-μέλη εκεί που διαπράττονται οι απάτες, αυτού του είδους η απάτη έχει διασυνοριακή διάσταση, πολύ συχνά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο και μόνο, και αποτελεσματική καταπολέμηση απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Στο άρθρο 5 ορίζεται η παρακίνηση, η υποβοήθηση και προσπάθεια, απόπειρα. Και πρέπει να προβληματιστούμε από αυτού. Ότι η απόπειρα δεν επεκτείνει στα ποινικά δικήματα που λέγονται στο 4, δεν καλύπτεται από αυτά. Μήπω υπάρχει δυνατότητα η απόπειρα, απόπειρα να θεωρείται ότι είναι τα ποινικά δικήματα που αναφέρονται στο άθρο 4. Παραγράφους 1, 2 και 3. Στο άρθρο 7 έχουμε κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα Υπάρχει αναφορά νομισματική στην παράγραφο 2, που να συζητηθεί το θέμα. Άρθρο 8, φυλάκιση, όρια φυλάκιση. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Ε, διάφορες υπεριστάσεις, δικές περιστάσεις, παραγραφή αδικημάτων μετά που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και αυτό είναι ένα θέμα προσυζήτηση το χρονοδιάγραμμα για την παραγραφή. Ελάχιστες κυρώσεις και αυτό είναι οριζόντιο ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε οι συγγητές και οι σκιώδεις και τέλος για τις τελικές διατάξεις το κεφάλαιο 4 συνεργασία μεταξύ κρατών μελών κατά την άποψή μου θα πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο την όλα Πρέπει να δίνει όλα τα κάτι μέλη τι πληροφορίε και να βοηθά τα κάτι μέλη να βοηθά στις έρευνες για να προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, και ούτω Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά. Να προσέξουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Έχουμε μόνο ένα χρόνο πριν το τέλο τη θητεία. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα θα δείξει τη δυνατότητα που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λειτουργήσει ως ε, νομοθέτη στον ποινικό τομέα. Είναι μια πρόκληση αυτή για μας. Πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό εξυπακούεται. Να συμπληρώσουμε το ποινικό νομικό πλαίσιο για την εμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων και να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μας νοιάζουν τα δικαιώματά τους. Χρησιμοποιήσουμε την αρχή της αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Έχουμε πολλή δουλειά. Εμείς οι συγγητές και σκιώδεις ας ακούσουμε τον υπεύθυνο συγητή της Επιτροπής ΚΟΝ, την εισηγήτρια μάλλον, την κυρία Γκρέσλε. Έχει το λόγο κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την κοινή συνεργασία γιατί η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού καθημερινά αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που ανακέπτουν και ε, και αν δεν μπορούμε να τα λύσουμε επειδή δεν έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο, ε, δεν είναι σωστό. Γι' αυτό θέλουμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια πολύ σωστή πρόταση. Η Κομισιόν Υπάρχει το άρθρο ε, 325 στη συνθήκη και θα ήθελα να επισέλθω στα προβλήματα εάν αλλάξει αυτή η νομική βάση. Θεωρώ ότι είναι προβληματικό και θα εμείνω σε αυτή τη θέση γιατί θεωρώ ότι είναι σφάλμα. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή της νομικής βάσης και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ποια είναι η στάση της νομικής υπηρεσίας. Η αλλαγή της νομικής βάσης δεν σημαίνει μόνο την τροχοπέδη αλλά θα έχουμε ένα δυνατότητα opt-out από τρεις χώρε μέλη και αυτό το opt-out θα σήμαινε ότι, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολύ δαπανηρές παράλληλες δομές. Γιατί για αυτές τις τρεις χώρες ε, αυτές οι υφιστάμενες δομές για την Europol και Eurojust θα πρέπει να παραμείνουν. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μια νέα δομή, αλλά θα υπάρχει και η παλαιά δομή. Και θα ήθελα να σε επισημάνω ότι κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δαπανηρό. Και θα ήθελα στη συνέχεια να θέσω ένα ερώτημα όσον αφορά τη δωροδοκία των βουλευτών μετά την αλλαγή της νομικής βάσης και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν πώς βλέπει αυτή την αλλαγή και θα ήθελα να διασφαλίσω τους συναδέλφους και τους συνηγητές ότι εγώ συγγήτρια της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού έχω μεγάλο ενδιαφέρον ή δυνατόν να υπάρξουν πολλές συζητήσεις με τους σκιώδες αλλά δεν θα ήθελα να ευνουχίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί η αλλαγή της νομικής βάσης θα έχει σαν αποτέλεσμα δυσκολίες που θα ανακύψουν μελλοντικά σε σημαντικά θέματα. Ε, δεν θα μπορέσουμε εμείς ε, να παρέμβουμε και θα μπορέσει το Συμβουλίο να περάσει τι δικές του θέσεις. Θα ήθελα να αναφέρω τώρα τη δική μας εργασία. Η οργάνωση με τη μεγαλύτερη εμπειρία ε, σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι η Όλαφ. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαστήριο βάσει του οποίο μπορούμε να μελετήσουμε τα προβλήματα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, εάν δεν προσέξουμε με την αρμόνιση. Ένα δίδαγμα το είναι και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη δικαιοσύνη στις χώρες μέλη. Και αυτή η Επιτροπή προσπαθεί να το πράξει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας ε, η Επιτροπή έχει θεσπίσει το scoreboard ε, και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα. Ε, και εάν η Επιτροπή μπορεί να μας ενημερώσει ποια είναι η πρακτική ποινικών διώξεων στις χώρες μέλη και ποια ελλείμματα υπάρχουν στην ποινική δίωξη στο επίπεδο των χωρών μελών, αυτό θα ήταν θετικό. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί στη βάση αυτή θα πρέπει να στηριχθούν η τροπολογία γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αρχή που να ισχύει για όλους, αλλά να υπάρχουν μέτρα τα οποία να συμπεριλαμβάνουν τα επιμέρους ελλείμματα των ε, διαφόρων ε, πρακτικών ποινική ε, δίωξης. Η Κομισιόν είπε ότι επειδή υπάρχουν ελλείμματα στο επίπεδο των χωρών μελών και γνωρίζουμε από τη δική μας εργασία πόσο διαφέρουν αυτές οι ελλείψεις μεταξύ των χωρών μελών, θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που να μας φωτίζουν σχετικά. Και θα ήθελα να μας πείτε ποιες θα είναι οι συνέπειες για την ένωμη τάξη των χωρών κρατών, εάν απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες μέλη ε, τα δικήματα εις βάρος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης εναρμονιστούν. Ε, και εφόσον υπάρχει δηλαδή άνηση αντιμετώπιση των ίδιων αδικημάτων ε, εντός της χώρας και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αυστηρότερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό να έχουμε ένα πρόγραμμα ώστε να αλλάξουν οι ένομες τάξεις των χωρών ε, μελών, ούτε ώστε να είναι συμβατέ μεταξύ του. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η συμβατότητα, θα ανακύψουν πάρα πολλά προβλήματα για να δούμε πώς γίνεται η δίωξη εκ μέρους της όλων αυτών ποινικών αδικημάτων, αυτό είναι εξαιρετικά ευρύ πεδίο και θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμες περισσότερες πληροφορίες. Και μετά από αυτές τις γενικές παρατηρήσεις θα ήθελα να έρθω στις λεπτομέρειες, οι οποίες επίσης αξίζουν την προσοχή μας. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο λέει ότι στο άρθρο 2 δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να την ε, συμπεριλάβουμε. Και θεωρώ ότι αυτές είναι θετικές ε, προτάσεις, και, αλλά και ίσως θα έπρεπε να κάνουμε σχετικά μια ακρόαση για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε στο άρθρο 3 ε, παράγραφος α, ε, απά της βάρος των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αρκεί η απλή χρήση ε, εσφαλμένων αριθμών, έστω και αν δεν έχουν ψήρει κάποια ζημία βάρος της Ένωσης. Αλλά θα πρέπει οι εισαγγελίε στο επίπεδο των χωρών μελών να, να δουν τι γίνεται με τις φορολογικές υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά. Ε, και στην Ελλάδα υπήρξε ε, μία περίπτωση απάτηση με τεράστιες επιπτώσεις. Λοιπόν, ε, το άρθρο 4. Εδώ θα πρέπει να τιμωρούνται οι χώρες μέλη όταν σε διαγωνισμούς τα ενεχόμενα μέρη πάλι δεν ε, χορηγούν όλες τις αναγκαίες εδώ πληροφορίες. Εδώ δηλαδή αρκεί η πρόθεση χωρίς να έχει επισύρει πραγματική ζημία. Ε, και το πώς ε, ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία ασχολούνται με την προκήρυξη διαγωνισμών ούτω ώστε να μην διασπείρονται εις βάρος τους εσφαλμένες ε, πληροφορίες ε, και αυτό είναι ένα έργο της Όλαφ. Θα πρέπει να ενισχυθούν και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρες μέλη και θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα. Το άρθρο 5 και 6 και άρθρο 7 ε, για την ε, ευθύνη των φυσικών προσώπων. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό κεφάλαιο γιατί εδώ εμπίπτουν και οι υπάλληλοι. Αυτή είναι αρμοδιότητα της Νομικής Επιτροπής και θα ήθελα ε, ρητά να συστήσω στους συναδέλφους της Νομικής Επιτροπής να δουν τον κανονισμό όπου οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι υπεύθυνοι και μπορούν ε, να ψήρουν ε, αδικήματα εδώ μέχρι φυλάξη ενός ε, έτους. Δεν ξέρω ούτε μια περίπτωση που να έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η διάταξη. Αλλά και όποτε το λέω μου λένε αλλά πρόκειται να το, συντομότερο δυνατόν να εφαρμοστεί. Εάν δούμε το αν θέλουμε να κάνουμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσωπικό συμβατό με αυτή τη διάταξη, ε, αυτό θα ήταν πραγματικά ευκταίο, γιατί ε, χρωστάμε στους υπαλλήλου ε, ασφάλεια δικαίου και πραγματικά θα ήμουν ευγνώμων του την Επιτροπή εάν πάρει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. το άρθρο 8 και 10 ε, ορίζουν τις ε, ελάχιστες ε, ποινές. Και αν δούμε πώς χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα των κυρώσεων και πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στις χώρες μέλη, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. συμπέρασμα. θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ενεχόμενων. Το νέο ευρωπαϊκό ε, δίκαιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το δίκαιο των χωρών μελών. Αλλιώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και θα προσκρούσει σοβαρά προβλήματα. Θα ήταν ε, καλό να μας πει ποια είναι η νομική βάση η οποία θα επιλέξει η Κομισιόν, γιατί η αλλαγή της νομικής βάσης σημαίνει ότι και η μελλοντική αυτή νομική βάση θα πρέπει να συμμορφωθεί με το εισφυστάμενο ε, πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much uh, to our Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκρέσλε. Καλωσορίζω το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, Τζοβάνι Γκέσλε Θέλουμε να ακούσουμε τώρα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα μόνο να τονίσω αυτό που είπε η συγγήτριά μας. Η αλλαγή της νομικής βάσης ε, από το 352 στο 83 πρέπει να διερευνηθεί και ε, ο συνάδελφος Λόπες Αγγιλάρ πιστεύει ότι θα ήταν σημαντικό να έχουμε μια κοινή αποτίμηση κινδύνου από τους νομικούς εμπειρογνώμονες και της δικής σας επιτροπής ε, με τρόπο ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς, ε, ποιες συνέπειες θα έχει αυτή η αλλαγή νομικής βάσης για μας. I suggest that προτείνω να ακούσουμε την άποψη όλων. Αυτό το ζήτημα συζητήθηκε εκτενέστατα ε, πρώτης και μεικτής συνεδρίας των δύο επιτροπών. Ε, έχουμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σχόλια τη κυρία Γκρέσλη εκτό μικρόφωνου. Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό της νομικής ε, βάσης για τη θέση του ε, Κοινοβουλίου υπεραμείνεται του άρθρου 83 αυτής της προσέγγισης. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τον εσωτερικό κανονισμό. Η κυρία Λεμπάη ήταν να τοποθετηθεί εξ ονόμων της Επιτροπής, αποχώρησε όμως. Ας ακούσουμε τον κύριο Κέσλερ, τον διευθυντή της Όλαφ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, έπρεπε να φύγει η κυρία Λεμπάη. Έχει μια άλλη πολύ σημαντική σύσκεψη και με άφησε, με παράτησε μόνο μου. Αυτά που θα σας πω ε, πάντως ε, είναι η κοινή τοποθέτησή μας με την κυρία Ντεμπάγε σε σχέση με την πρόταση οδηγίας για τις δύο υπηρεσίες Όλαφ και ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, είναι η κοινή θέση των δύο συναρμοδίων ε, υπηρεσιών. Αυτή ήταν ανέκαθεν η θέση τους. Δεν έχουμε αλλάξει θέση. Η κυρία Λεμπάη ε, μας άφησε τις γραπτές παρατηρήσεις της και είναι στη διάθεση των μελών της Επιτροπής. Uh, let me underline. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το φάκελο να είναι ισχυρή η παρουσία του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και ιδίω η Επιτροπή Κοντ ήταν μία από τις ε, κινητήριες δυνάμεις ε, για την προστασία του σημερινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Αυτή τώρα η οδηγία πώς στόχο έχει να καλύψει σε μεγάλο μέρος ε, επιμέρους στοιχεία του πρώην τρίτου πυλώνα, PFI, ε, τη σύμβαση του 99 και το πρωτόκολλο της ε, διαφθοράς ε, του 96 PFI και το δεύτερο πρωτόκολλο του 97. Δεν αρχίζουμε δηλαδή από το μηδέν. Αυτή η οδηγία είναι το δεύτερο σημαντικότερο βήμα προς την σε εισαγωγικά λισαβονοποίηση αυτών που συνέβαιναν βάσει συμβάσεων και πρωτοκόλλων ε, συμβάσεων. Η λισαβονοποίηση αυτού του ζητήματος ε, ε, καθίσταται απαραίτητη μεταξύ άλλων με στόχο για να κατοχυρωθεί στη συνήθινομοθετική νομοθετική διαδικασία ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Το πρωτογενές μέσο, οι συμβάσεις, εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη μόνο, από το Συμβούλιο και κατατίθεντο προς διαβούλευση αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο. Είναι η χρυσή ευκαιρία ε, σήμερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να διαδραματίσει κέριο ρόλο σε αυτόν τον τομέα κατά τη διαστολή με το παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε την οδό της λισαβονοποίησης. Και το άρθρο 325 της συνθήκης χρησιμοποιείται ως νομική βάση γιατί αυτό είναι το ενδεδειγμένο μέσο ώστε να αξιοποιήσει το Κοινοβούλιο αυτή τη νομική δυνατότητα και να εμπλακεί πλήρως, ε, ε, να είναι εταίρος σε αυτή την άσκηση. Ισότιμος εντός του Συμβουλίου σε αυτή την άσκηση. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν συζητήσει σε πολλά φόρα το, την οδηγία αυτή ε, και ε, ξαναλέω ότι δεν αρχίζουμε από το μηδέν. Το κεκτημένο που έχουμε αποκτήσει χάρη στα προηγούμενα μέσα είναι το πρότυπο της ελάχιστης προστασίας που έχουν μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, Γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει κάποιοι ε, να χρησιμοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για να αποσταθεροποιήσουν ακριβώς αυτό το κεκτημένο που κληρονομούμε από τα προηγούμενα ε, εργαλεία και από τις κείμενες συμβάσεις. Είναι ζωτική σημασία ο ρόλο του Κοινοβουλίου για αυτό το ζήτημα για να μην αποδυναμωθεί το κεκτημένο. Το αντίθετο θα πρέπει να επιτύχουμε ε, υψηλότερο επίπεδο ε, εναρμονισμένων και επικαιροποιημένων προτύπων ε, στον τομέα αυτό. some critical points. Κάποια πολύ βασικά σημεία θα ήθελα να εκθέσω ε, κριτικά για την κρίσιμη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη σκοπιά της Όλαφ. From the key of... Το κεκτημένο από τη σύμβαση του 1995 και ε, των πρωτοκόλων της σύμβασης σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής κυρίως του νομοθετήματος και με τον ορισμό της απάτης και θα ήθελα να αγγίξω και κάποιες άλλες διαστάσεις του ζητήματος. Ας αρχίσουμε όμως από το πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να είναι η ευρύτε, το ευρύτερο δυνατό για να καλύπτονται όλα τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες. Ε, ανεξαρτήτως μέσων ε, ε, δαπανών. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε καλύτερο πεδίο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Όλα το σύνολο των εσόδων που προβλέπονται στην απόφαση για τα ίδια μέσα, τα έσοδα από το ΦΠΑ, όλα, όλα τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτονται. Επίσης, στην περίπτωση λαθρεμπορίου των τσιγάρων παραδείγματος παραδείγματο χαρή, η απώλεια, τα διαφυγόντα έσοδα ε, επιβαρύνουν όχι μόνο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους φορολογούμενους ε, ε, των κρατών μελών που θα πρέπει να καλύψουν το κενό στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αναφέρθηκε ήδη από τον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ το ζήτημα του ΦΠΑ. Είναι προφανές για μας ότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί διότι συνιστά οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και μείζον πόρος για την ε, Ένωση. Ε, είναι απαραίτητο να διευρύνουμε το πεδίο και να προστατεύσουμε τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ε, τα χρήματα των φορολογουμένων και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο πεδίο αρμοδιοτήτων για το Γραφείο της Εισαγγελίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε από την σκοπιά της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ο ορισμός της απάτης. Ένα σημαντικό και εκτιμένο της ε, προηγούμενης αλλά και κείμενης νομοθεσίας, των συμβάσεων δηλαδή, που ισχύουν στον τομέα αυτό είναι το εξής. Και να πω παρενθετικά ότι δεν θα θέλαμε ο ορισμός στον οποίο έχουμε καταλήξει η δυνάμη του ε, ισχύοντος ε, πρωτόκολλου να περιοριστεί, διότι αν περιορίζαμε το πεδίο του ορισμού της απάτης, αυτό θα ήταν επιζήμιο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την προστασία αυτού. Το αντίθετο. Θα πρέπει να επεκταθεί να διευρυνθεί ο ορισμός για να καλύψει κάποια δεδομένα, κάποια επιμέρους στοιχεία που τα τελευταία δέκα χρόνια αποδεδειγμένα είναι επιζήμια προς τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε αξιόπινες πράξεις όπως απάτε στους ε, διαγωνισμούς για κρατικές προμήθειες. Στην πράξη η Όλαφ έχει καταδείξει ότι ε, αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ε, παρόλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της απάτης, παρότι είναι επιζήμιο για τα συμφέροντα της Ένωσης και γι' αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί στην, στο σχέδιο οδηγίας. Τέλος, το θέμα της παραγραφής των αξιόπινων πράξεων. Ε, καταθέσαμε αυτή την πρόταση για να εναρμονίσουμε την περίοδο παραγραφής για τα, ε, τις αξιόπινες πράξεις που προβλέπονται στην οδηγία. Ελάχιστος χρόνος ορίζεται στα πέντε χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εναρμονίσουμε τις περιόδους παραγραφής σε όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η δίωξη από τις εθνικές αρμόδιες αρχές και να επιτύχουμε την καταδίκη των ε, ενόχων. Δεν διώκονται κάποια δικήματα ακριβώς ε, λόγω της εκπνοής της περίοδου παραγραφής ε, που διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό από κράτο σε κράτο αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ένας ε, βασικός λόγος ανησυχίας και ατιμορρησίας αυτών των αξιόπινων πράξεων παρά τη διακύμανση της ε, περίοδου καταλαβαίνετε ότι συνιστά εθνική αρμοδιότητα και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως προς την περίοδο παραγραφής. Είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε θα πρέπει να διευθετήσουμε, εξού και η πρότασή μας ε, προς εναρμόνιση. Ταυτόχρονα είδαμε ότι οι υπέτειοι εύκολα μπορούν να επιλέξουν σε ποιο κράτος μέλος θα έχουν τον τραπεζικό λογαριασμό, πού θα υπογράψουν ε, τις ε, συμβάσεις, ε, ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο παραγράφησε Στην πράξη αυτό εξισούται με ατιμορρησία και ή με μεγάλη δυνατότητα να πετύχει κανείς τον απότερο στόχο που είναι η ατιμορρησία. Γι' αυτό και προτείνουμε την αλλαγή της νομικής βάσης. Προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 325 και όλος ιδιαίτερο στο εδάφιο 4 ε, είναι μια πολύ ειδική διάταξη, χάρη στην οποία μπορούν να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των οικονομικών σφαιρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της απάτης ε, ε, μέσω από αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα. Επινικές διαδικασίες και ποινικέ κυρώσεις μπορούν να προβλεφθούν μάλλον χάρη σε αυτές τις διατάξεις. Αυτό είναι ο στόχο τη νομική βάση και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Επιβεβαιώθηκε η ερμηνεία μα από πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ποινική υπόθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πλήρη επίγνωση του ότι είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο το ζήτημα και συζητείται επί μακρόν και στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και προσβλέπω στην εμβάνθυνση του ζητήματος ε, στις μελλοντικέ μας συζητήσει σχετικά με τη χρήση αυτού του ε, νομικού εργαλείου που ε, θα συνιστά τη νομική βάση για αυτή τόσο σημαντική οδηγία. Ο Πρόεδρος, κ. Λόπες σας υπενθυμίζω ότι στις 10 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και τα μέλη της Επιτροπής ΚΟΝ σίγουρα έχουν και ε, ανηλυμένες υποχρεώσεις. Σας παρακαλώ ως εκ τούτου να είναι συντομότατες παρεμβάσεις διότι έχουμε τον εκπρόσωπο της Ιρλανδικής Προεδρίας ακόμη ε, και άλλα δύο μέλη της Επιτροπής που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών. Παρακαλώ, ναι, ναι, η εκπρόσωπος της Ιρλανδικής ε, Προεδρίας. Σας ακούμε. Uh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε τη Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, εξότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνάδελφοι, θα είμαι συντομότατη. Όπω ήδη αναφέρθηκε, ελπίζουμε ότι στο Συμβούλιο σε δύο εβδομάδε περίπου δικαιοσύνη και εσωτερικών θα έχουμε συμπεφωνημένη γενική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σημαντικό για όλους τους παρόντες να σημειώσουν ότι η γενική προσέγγιση συμφωνήθηκε επί της νομικής βάσεως του 832 αυτή ήταν η θέση του Συμβουλίου και υπήρχε μια πολύ ισχυρή μεγάλη πλειοψηφία που υποστηρίζει τη νομική βάση αυτή ε, και αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Η βάση είναι το 83-2, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ε, είχαμε εξαιρέσει κάποια πράγματα από τον ορισμό ε, και το θέμα των ελάχιστων κυρώσεων ήταν πάρα πολύ επίμαχο ζήτημα και είναι μια κόκκινη γραμμή για τα κράτη-μέλη αυτή. Το θέμα των ελαχίστων κυρώσεων στο συγκεκριμένο μέσο ε, δεν υφίσταται στην γενική προσέγγιση. Άλλα θέματα προφανώς έχουν αλλάξει. Σε άλλους τομείς είδαμε να υπάρχουν διαγραφές από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα των κρατικών προμηθειών, των δημοσίων προμηθειών. Ειδεμή, ελπίζουμε το συμπεφωνημένο κείμενο που συμφωνήθηκε σε επίπεδο ομάδας εργασία να εγκριθεί ε, τις επόμενες ε, δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δήλωση που έκανε η Ιρλανδική Προεδρία. Λοιπόν, τα μέλη θέλουν να πάρουν το λόγο. Σας υπενθυμίζω ε, ότι θα έπρεπε ίσως να είσαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ο κύριος Ντένις Δε Γιόγκ, που ήταν εισηγητής υπεύθυνο για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το ποινικό δίκαιο, Κύριε Ντε Γιόγκ, ο κύριος Ντε Γιόγκ, α, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θέλουμε να έχουμε συνέπεια. Και γι' αυτό θα ακολουθήσω λογική προσέγγιση. Και μάλιστα γι' αυτό απογοητεύτηκα με την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα για την νομική βάση. Είχαμε το άρθρο 83.2 που το ανέφερα και στην έκθεσή μου σαν βάση για μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Να εξετάζεται σαν πακέτο και όχι κατακαιρματισμένη αντιμετώπιση σε κάθε επιτροπή. και η ιδέα του Κοινοβουλίου όταν υιοθέτησα την έκθεσή μου ήταν να ακολουθήσουμε πιο συνεπή οριζόντια προσέγγιση. Νομική βάση. Θεωρώ ότι δεν βοηθά η πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Κατανοώ αυτό που είπε η Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη-μέλη. Αν διατηρήσουμε το 83, έχουμε τουλάχιστον την οριζόντια προσέγγιση. Και τι σημαντικότερο, υπάρχουν προτάσεις εδώ, σε αυτό το τομέα, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων για ελάχιστε κυρώσει για μεγαλύτερη εναρμόνιση των ε, ε, ορίων παραγραφής και των ορίων γενικά και αυτά θα πρέπει να συζητηθούν οριζόντια όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Δεν μπορεί κανείς να θεσπίσει ελάχιστες κυρώσεις από τη μια και παραποίηση του ευρώ από την άλλη, παραχάραξη του ευρώ και τώρα στην παραποίηση, στην ε, υπονόμηση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εάν θέλουμε ελάχιστα, ελάχιστες κυρώσεις θα πρέπει να εισαχθούν αυτές σε όλο το σύστημα του ποινικού δικαίου και θέλουμε να έχουμε μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελάχιστες κυρώσεις. Ρώτησε την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ στην Επιτροπή Λίμπε και είπε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δείτε κάτι μέλη πιθανότατα δεν το δεχτούν αυτό. Αλλά είναι εσφαλμένη η προσέγγιση αυτή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, βλέπει κανείς το υπόβαθρο τη μάχη που γίνεται μεταξύ Όλαφ και Eurojust. Η επιλογή της νομικής βάσης, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινείται προς την κατεύθυνση της Όλαφ να είναι η βάση για τον ε, Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αν επιλεγεί το άρθρο 83 παράγραφος 2, κινείται περισσότερο προς την κατεύθυνση του Eurojust αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Στην ΚΟΝΤ, μετά από αυτή τη συνεδρίαση, θα διεξαχθεί συζήτηση όσον αφορά τη λειτουργία τη Όλαφ, στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τον πίτρο Νταλή. Διάβασα όλη την τεκμηρίωση και συγκλονίστηκα από τη συμπεριφορά τη Όλαφ σε αυτή την έρευνα. Παραβάσατε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, του κατηγορούμενου και με βάση αυτό το ιστορικό θα δίσταζα πολύ στο να εμπιστευτώ την Όλαφ σαν ε, την αρχή, σαν τη βάση της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάνν Άλμπρεχτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους που μας δίνουν το χρόνο για την σημαντική αυτή συζήτηση. Συμφωνούμε όλοι ότι η καταπολέμηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο να αντιμετωπιστεί. Έχω και εγώ κάποιες αμφιβολίες, όπως και συνάδελφος, όσον αφορά τη νομική βάση. Μιλάμε για τον ευαίσθητο τομέα του ποινικού δικαίου είναι πολύ σημαντικός τομέας που αφορά το συνταγματικό δίκαιο των κρατών μελών και αναφερόμαστε σε ένα τομέα που όσον αφορά την ευρωπαϊκή διαμόρφωση πολιτικής είναι στο μέσο όπου η επικουρικότητα και οι αρχές και οι κανόνες που αναφέρονται σε ισορροπημένη προσέγγιση στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και στα ανθρώπινα δικαιώματα του Δικαστηρίου του Στρασβούργου παίζουν ρόλο. Είναι πολύ ευαίσθητο τομέα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριζοντίω. Χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση. Οπότε κατανοώ το επιχείρημα. Εν γέννη πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 83 για την αρμόνιση του ποινικού δικαίου να θεσπίσουμε ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, να έχουμε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τον ευαίσθητο τομέα. Δεν αρνούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να βάσουμε τα μέτρα του ποινικού δικαίου, κυρίως εναρμονισμένες κυρώσεις επί του άθου 325, αλλά από πολιτική σκοπιά αυτό δεν θα ήταν πολύ συνετό, διότι όπως ήδη είδαμε, η συζήτηση για την Όλαφ και τα ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά το δίκαιο που θα εφαρμοστεί, αρχές, θεμελιώδεις αρχές, βλέπουμε από όλα αυτά ότι χρειάζεται νέα προσέγγιση όσον αφορά τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις διάφορες ποινικέ υποθέσεις στο ποινικό δίκαιο, οπότε θα σας καλούσα να βαθίσουμε τις νομικές πράξεις στο άθρο 83, παρόλο που βλέπω ότι βέβαια για το Κοινοβούλιο αυτό συνεπάγεται συνέπειες και συνεπάγεται συνέπειες και για τις νομικές πράξεις. Θα πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε εντό τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχουμε μεγαλύτερε δυνατότητε εναρμόνιση του ποινικού δικαίου, περισσότερε δυνατότητε να θεσπίσουμε νομικές ε, διαδικασίες και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το ζήτημα μέχρι να έχουμε τις συνθήκες της ε, χρησιμοποιήσαμε αρμοδιότητε απέναντι από τι διατάξει τη συνθήκη, αλλά έχουμε λέξει σπεσιάλη ειδικό δίκαιο με τη νέα συνθήκη και όπως λέει η νομική επιτροπή και εγώ θα ήθελα να διαλέξουμε ω νομική βάση τα 83. Αλλά θα σας παρότρινα να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζεται εναρμόνιση στον τομέα. Πρέπει να συνεχιστεί η εναρμόνιση και καλό και το Συμβούλιο να μην μπλοκάρει την πρόταση για τον εισαγγελέα, τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε κοινέ αρχές, εναρμόνιση ποινικού δικαίου και χτες τελείωσαν οι τριμερείς διάλογοι για την πρόσβαση στα αρχεία των νομικών. Είναι η προϋπόθεση αυτή για την αρμόνιση του ποινικού δικαίου και πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί και να ακολουθήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν. Είναι σημαντικό να είναι συνεκτική προσέγγιση και στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να συζητήσουμε το ποινικό δίκαιο εν γέννη. Πού το τοποθετούμε όσον αφορά τις διάφορες αρμοδιότητες που έχουν οι επιτροπές. Έχουμε μόνο 5 ή 7 λεπτά και υπάρχουν τρεις ε, ε, βουλευτές που θέλουν να παρέμβουν. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ε, συγγνώμη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το ερώτημά μου, λέει η κυρία Γκρέσλε. Συγγνώμη, καταρχήν ε, ο κύριος Γιακολίνο και μετά θα επανέλθουμε σε εσάς σου συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναφισβήτητα, Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις ε, παρεμβάσεις, στοιχεία προς προβληματισμό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν ξέρουν πρώτα απ' όλα της κυρία Νταβέλ την άποψη, διότι έπρεπε να αποχωρήσει από τη συζήτηση. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την κυρία Ντεβάλε. Από αυτά που υπόθηκαν, διαφαίνεται ότι το Συμβούλιο στο πεδίο εφαρμογή της οδηγία δεν θέλει να συμπεριλάβει τον ΦΠΑ που η Γενική Διευθύντρια Κέσλερ ε, θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή. Οι συγητέ σε αυτή τη φάση διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει το πεδίο εφαρμογή πρέπει να είναι το ευρύτερο δυνατό. Η καταπολέμηση των απατών γίνεται μέσω στεναρής δικαστικής και αστυνομική συνεργασίας που εδράζεται επί εμπιστοσύνης των κρατών μελών αλλά και μέσω πιο στενής επαφής και διάδοσης των πληροφοριών. Πέρα από την νομική βάση που θα καθοριστεί. Σίγουρα όλα αυτά ε, υπονομεύουν, οι απάτες υπονομεύουν την νόμιμη οικονομία και έχει και κοινωνικές συνέπειες η απάτη. Διότι μειώνται τα έσοδα μέσω των, λόγω των απατών. Κύριε Πρόεδρε, σαν εισηγητής, κάντε ό,τι μπορείτε και σαν πρόεδρος Επιτροπής, ούτως ώστε στο Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε μια πρόταση για την ε, εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Περιμέναμε να γίνει αυτό τον Ιούνιο, έχουμε καθυστερήσει όμω πολύ. Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματο και πολύ συχνά σε αυτά τα πλαίσια των συζητήσεων πρέπει, ε, συμμετέχει το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι συγητές με τους διάφορους φορείς μαζί με την Όλαφ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα του πεδίου εφαρμογής δεν θα υπάρξουν ελάχιστε κυρώσει. Το μαθαίνουμε τώρα, γιατί δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη υπό την ελάχιστον κυρώσεων. Και για τι απάτε στο ΦΠΑ έχουμε μεγάλε δυσκολίε. Κλείνω. Και λέω ότι είναι εξίσου σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε μέτρα που αφορούν, ε, αφορούν την, την κατάσχεση των παρανόμως ε, συλλεχθέντων εσόδων. Τέτοιες κατασχέσεις αυτό το στοιχείο ενεργητικού από παράνομε πράξει θα μπορούσαν να βοηθήσουν να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση αυτή τη ε, ε, οδηγία, η εφαρμογή τη οδηγία. Ο κ. Μπαλσίτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου άποψη για τα θέματα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Όλαφ είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερευνά φαινόμενα απάτηση ε, και η Όλαφ δεν είναι όμως σε θέση να λάβει επαρκείς πληροφορίες από τις χώρες μέλη και ποιες ποινές ε, επιβάλλονται. Κατά την άποψή μου κάτι τέτοιο δεν είναι παραδεκτό και θα πρέπει να περιλάβουμε αυτό το στοιχείο στην λόγο οδηγία. Η κυρία Γκρέσλεν, συντομία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμπενθυμίσω όμως τη δική μου ερώτηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Συμβούλιο έχει ήδη ε, καταπατήσει τη νομική ε, βάση, ε, καταθρηματίσει τη νομική βάση. Ε, και εμείς τελικά το στηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι χρειαζόμαστε πληροφορίες για την ε, ε, πρακτική των ποινικών διώξεων στο επίπεδο των χωρών μελών και τις ενδεχόμενες ελλείψεις. Ε, αν δεν επικεντρωθούμε στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα πάνε στραβά τα πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε ε, το πρώτο βήμα πριν από το τρίτο βήμα. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα θα δούμε όταν έρθει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδυναμωθούμε ευθύ εξ αρχή, γιατί δεν έχουμε το πρώτο, την πρώτη, το πρώτο βήμα, δεν κάνουμε το πρώτο βήμα, θα αποτύχουμε. Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι διευκρινίσαμε κάποια πράγματα ε, πριν ε, ολοκληρώσουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Κάποια λόγια από τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Θα ήθελα να πω εν συντομία ότι συμφωνώ απολύτως με την κυρία Γκρέσλε στα όσα είπε στην τελευταία της παρέμβαση. Δεν θα ήθελα εδώ να προσθέσω τίποτα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και έχουμε τη νομική βάση να το πράξουμε. Ε, και για το Κοινοβούλιο αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία. Από την άλλη, η νομική βάση δεν ε, σχετίζεται με την όλαφη ή με τη Eurojust κατά κανένα τρόπο. Κανείς μπορεί να αγαπάει την Όλαφ ή να τη μισεί, το ίδιο τη Eurojust ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτά δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτή η πρόταση έχει σαν σκοπό να εναρμονίσει την υφιστάμενη νομοθεσία στις χώρες μέλη, η οποία μέχρι σήμερα δεν είναι ενημερωμένη ε, εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και ανοίγει την πόρτα σε φαινόμενα απάτης. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Γκρέσλε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ε, Επιτροπής ε, Προπολογισμού. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να βελτιώσουμε την ανταλλαγή απόψεων και συζήτησα με τον συνάδελφο κ. Γιλάρ ότι θα είχε νόημα ίσως να οργανώσουμε το συντομότερο μία ακρόαση με τους επιτρόπους που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Ε, θα θέλαμε να ευχαριστούμε τον συμπρόεδρο κύριο Τόιερ και όλους τους ε, συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ε, το άρθρο 325 ισχύει, αλλά επίσης και το άρθρο 83 και το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να προσπαθήσει μια συμφωνία. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια συζήτηση όπου οι συγητές και οι σκιώδεις να διερευνήσουν όλες αυτές τις δυνατότητες και ελπίζουμε ότι αυτή η εντολή θα είναι χρήσιμη ούτω ώστε να δείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει, είναι στο αντάξιο στην, στο έργο, στην αποστολή της ε, νομοθεσίας.